Okay, friends. Try to find yours. Παρακαλώ προσπαθήστε να καθίσετε Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Μπορείτε να βάλετε την κάρτα ψηφοφορία σας ε, στο μηχάνημα για να αρχίσουμε την ψηφοφορία με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, την κινητοποίησή του για την Good Year. Είναι ε, ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Sorry. Yes, and Πέρας ψηφοφορίας. And it's 40 uh, votes. 44 υπέρ. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία με τις συμβιβαστικές. Συμβιβαστική L, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην αλλακτική συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ηλεκτρονικός. Έναρξη ψηφοφορίας. Υπάρχει ένας υπεράριθμος. Από το ΕΛΚ. Does it work when I when I? How do you not when closed? I don't know. Is it just there? I. Sorry for that. Uh, yes. It... Συγγνώμη, λοιπόν, απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 99 υπέρ. Κατά. Έλεγχος της 99. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛ ψήφισε. I can't see the figures. No, no. no. I, I don't... And it's, it's carried with one vote. Εγκρίνεται. Όχι. Συγγνώμη, υπάρχει ένας αδικατοπτρισμός με το φως και δεν βλέπω καλά. Εντάξει, εγκρίνεται. Συμπεβαστική M, υπέρ. Απορρίπτεται, απορρίπτεται, συγγνώμη. Συμπεβαστική M, υπέρ. Κατά. Έλεγχος της M. Εγκρίνεται. 92. Όχι. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική N υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική O υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική π υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος, έλεγχος, έλεγχος της συμβιβαστικής R. And the vote is open. The vote is now... Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εκατόν υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος της 128. Πέρας. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Uh, we go to amendment 135 υπέρ. Κατά. Πρέπει να την ελέγξουμε την 135. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 27 προς 21. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 145 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά έλεγχο του δεύτερου τμήματος της 145 έναρξη ψηφοφορίας πέρας απορρίπτεται 146 όχι 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εναλλακτική συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρας της ψηφοφορίας 24 προς 19 απορρίπτεται Τροπολογία τώρα 152 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ α όχι πηγαίνουμε στην 157 απευθεία συγγνώμη 157 λοιπόν υπέρ κατά έλεγχος της 157 έναρξη ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. 26 προς 20. 158 υπέρ. Κατά αποχές. Να την ελέγξουμε καλύτερα την 158. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται με 26 ψήφους. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 όχι, λάθος. 167 λέει πρόεδρος με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Y, υπέρ, κατά, έλεγχος τη συμβιβαστική Y. Έναρξη ψηφοφορίας, πέρας, Εγκρίνεται με 24 ψήφους. Πηγαίνουμε λοιπόν στην επόμενη σελίδα, στην 180 τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AA, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 190 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 247 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 191 είναι μια ψηφοφορία με ονομαστική κλίση την οποία ζήτησαν οι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Έναρξη λοιπόν ψηφοφορίας για την 191. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 25 ψήφους. Τροπολογία 194. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Της 194. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρασα. Εντάξει. Εγκρίνεται. με 30 ψήφους. Συμβιβαστική AC. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Τις 202. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με 28 ψήφους. Τροπολογία 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AD υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AE υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά Έλεγχος της 223. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική AG υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται Συμφιβαστική AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 230 υπέρ κατά έλεγχος της τροπολογίας 230 έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται με 29 ψήφους. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AI ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ε, συγγνώμη, 237 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AJ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 244 υπέρ κατά αποχές νομίζω να ελέγξουμε τη 244 έναρξη ψηφοφορίας Πέρας. Απορρίπτεται. Με 20 ψήφου. 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΕΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 255. Πρώτο τμήμα. Α, συγγνώμη, δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα της 255 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος έλεγχος του δεύτερου τμήματος τροπολογίας 255 έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται με 25 ψήφους τροπολογία 256 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Έλεγχος του δεύτερου τμήματος της 256. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Με διαφορά τριών ψήφων. Καλτ 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 10 συγγνώμη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλτ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα πάμε στις αναφορές. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ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 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε λογικέ σκέψεις. Συμβιβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά Και επαληθεύουμε για να βεβαιωθούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 27 ψήφι κατά 20 υπέρ. A ε, συμβαστική A υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ή ε υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 57 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την 57 άρχεται πέρας εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ 18 κατά G συμβιβαστική G υπέρ κατά επαληθεύουμε μια ναι, και δεν σηκώνεται αρκετά τα χέρια συμβαστική G λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται ομόφωνα σχεδόν 42 ψήφοι υπέρ παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η κάπα συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές συμβαστική είναι από την αρχή συμβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ευχαριστώ Συμβαστική H ή τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, Ι, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα τέσσερα υπέρ κατά και επαληθεύουμε. Εβδομήντα τέσσερα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται με τέσσερις ψήφους διαφορά. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. J, συμβαστική J, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΙΑ συμβαστική ΙΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απερίφθη λέω εγώ αλλά ας επαληθεύσουμε 83 Πέρα της ψηφοφορίας και εγκρίνεται 29 ψήφι υπέρ 18 κατά. 86 τώρα υπέρ κατά. Αποχές και επαληθεύουμε την 86. Αρχίζει η ψηφοφορία στην 86, πέρα της ψηφοφορίας. και εγκρίνεται 27 υπέρ, 21 κατά. 87 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Τη ψηφοφορία για το σχέδιο εκθέσεω όπω τροποποιήθηκε. Εγκρίνεται λοιπόν 24 ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά, 14 αποχέ. Και ευχαριστούμε τον εισηγητή. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο. Το θέμα τώρα της απάντησής μας προς το Συμβούλιο και ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προχωρώ στην τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ, κατά αποχές. Επαληθεύουμε την τροπολογία υπαριθμών 1, αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν 25 προς 22. Τροπολογία 2 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε νομίζω. Τροπολογία 2. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα τα μηχανήματα. Σας παρακαλώ να επαληθεύσουμε, να επαναλάβουμε την επαληθεύση για την τροπολογία υπαριθμών 2. Τώρα λοιπόν κλείνει οριστικά η ψηφοφορία και εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ 19 κατά. 7. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Οχτώ υπέρ κατά χέσα... και επαληθεύουμε την 8 πέρας 26 ψήφι σχέδιο προφορικής ε, ε, ερώτησης ονομαστικά όπως είπαμε και πέρα της ψηφοφορίας. Σεραντοχτώ ψήφι υπέρ, κανένα μία ψήφος κατά, ψήφισμα. Κυρία Ράνκη, έχεις στήσει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το ψήφισμα εδώ ε, είδε χτες αργά το βράδυ την τελευταία στιγμή συμβαστικές τροπολογίες. Ήταν πολύ δύσκολο για μας, αλλά και για άλλους συναδέλφους να ε, προετοιμαστούμε, να διαβάσουμε σωστά τις συμβαστικές τροπολογίες και να επιλέξουμε στάσεις στην ψηφοφορία. Γι' αυτό θα σας παρακολούσα να αναβληθεί για λίγο η ψηφοφορία, να μπορέσουμε να μελετήσουμε εις βάθος τις τροπολογίες. Ξέρω ότι στηρίζονται σε τροπολογίες που είχαμε στο παρελθόν καταθέσει, αλλά επειδή έχει γίνει συγχώνευση περισσότερων της μιας τροπολογιών, θα ήθελα να δοθεί λίγος χρόνος Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για τις ομάδες να μπορούν να μελετούν τις τροπολογίες τις συμβαστικές και όταν αυτές κατατίθενται με τόση καθυστέρηση είναι αδύνατον. Δηλαδή τι λέτε να μην ε, ψηφίσουμε τώρα. Σας παρακαλώ να γίνει ψηφοφορία με ερώτημα την αναβολή για την προσεχή δυνατότητα ψηφοφορίας του θέματος αυτού. Ωραία λοιπόν λέει ο Πρόεδρος. Ποιος θέλει την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας. Παρακαλώ. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την 23 παρακαλώ 23. Πέρας της τώρα. Και απερίφθη. 64 σε τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές απερίφθη Συμβιβαστική 66, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά. Εγκρίνεται άκαλα να επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Έχουμε έναν ε, περισσευούμενο και από το ΕΡΚ και από τους αλληστές Δημοκράτες. Παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας και απεριφθεί. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη επαληθεύουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα και αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ένας περισσευμένος από το ΕΛΚ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη δηλαδή. Τρίτο τμήμα. Α, καταπίπτει το τρίτο τμήμα. 70, τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Σε τμήματα η 72, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές. Λέω ότι απερίφθημένα, αλλά ας το επαληθεύσουμε όπως και να έχει. Δεύτερο τμήμα λοιπόν. Πέρας. 26 ψήφι κατά και απεριευθεί. 24 τώρα, συμβαστική 24 υπέρ κατά. Αποχές. Απεριευθεί. 73 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την 78 αρχίζει πέρας και απερίφθη 26 ψήφοι κατά 79 υπέρ κατά εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να επαληθεύσουμε την 81 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 28 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται, 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ κατά ε, την 84 πέρας Εγκρίνεται 23 υπέρ 19 κατά. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά και επαληθεύουμε πέρας 27.92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 όχι 111 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την 111 πέρας προφορίας. Με 27 ψήφους εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ συμβαστική 28 κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και επαληθεύουμε την 148 πέρας απερίφθη Απερίφθη. Με τρεις ψήφους η φορά. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά και να επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα της 156 πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη με 34 ψήφους κατά. 157 παρακαλώ υπέρ. 157 υπέρ. Κατά αποχές απεριφθή Θα επαληθεύσουμε 157. Αρχιετή ψηφοφορία και πέρας. Και εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. 158 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά επαληθεύουμε την 160 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ, 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται 175 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά. Αποχές απερίφθη και επαληθεύουμε την 177. Πέρας. Και απερίφθη. 178 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 183 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε την 183 πέρας εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ 184 υπέρ κατά και επαληθεύουμε μα γιατί πολύ λίγοι σηκώνετε τα χέρια σας Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη με τέσσερις ψήφους διαφορά. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε την 189 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ 190 υπέρ κατά αποχές επερίφθη 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 194 υπέρ κατά αποχές απερίφθη και πάμε στις αιτιολογικές αναφορές νούμερο ε, πρώτη, αναφο... πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτη υπέρ κατά αποχές απερίφθη αιτιολογικές σκέψεις συμβαστική πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά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 και περιφθεί με μία ψήφο 25 υπέρ. Και επαληθεύουμε την 25 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 27 ψήφοι υπέρ. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Επαληθεύουμε την 26, πέρας της ψηφοφορίας. Έχει έναν περισφομενό το ΕΛΚ. Τώρα θα δούμε το αποτέλεσμα. Όχι. Τώρα ναι. Και απερίφθη. Συγγνώμη, απερίφθη, απερίφθη. Συμβαστική 21 υπέρ. Μ' αρέσει φαίνεται το κόκκινο, γι' αυτό μπερδεύομαι και ο λέω εγκρίθηκε, ενώ έχει απορριφθεί. 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται λέω. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Επαληθεύουμε την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 35 υπέρ κατά αποχές απερίφθη όχι θα το επαληθέψουμε νομίζω ότι έχει κρυθεί. Πέρα τη προφορία εγκρίνεται με 28 ψήφου υπέρ. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Σαράντα τρία υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 44 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 60 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και δεύτερο υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε. 42 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά και 2 αποχές και συγχαρητήρια στους εισηγητές για την πολύ καλή δουλειά. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ψηφορία, Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Κάρτα και ξεκινάμε με τις τροπολογίες 16 και 17 που θα ψηφιστούν σε μία τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. κατά έλεγχος, επαλήθευση μάλλον, επαλήθευση της ψηφοφορίας. Παρακαλώ ψηφίζετε και έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία με 29 ψήφους. σημαίνει ότι περνάμε απευθείας στην τελική ψηφοφορία γιατί με βάση αυτό που ψηφίσαμε περνάμε απευθείας στην τελική ψηφοφορία για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Περνάμε δηλαδή σελίδα υπεριθμών 11 και Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Can Μήπως μπορείτε λιγάκι να επαναλάβετε αυτά που είπατε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έχετε την καλοσύνη να επαναλάβετε. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ίσως να μην το λέω καλά στα αγγλικά αλλά ε, αναφέρουμε στην τελική ψηφοφορία που αναφέρεται στη σελίδα υπαριθμών 11 ε, και θα ψηφίσουμε για, την, ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ και έληξε η ψηφοφορία. and it's carried by 28 votes. Thank you, Madam Harkin. Uh, Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για την ε, πρόταση για οδηγία σχετικά με την ηλεκτρονική κάρτα. Οδηγία για την ηλεκτρονική κάρτα. Ψηφίζουμε για τι ε, τροπολογίε υπαριθμών 17 και 18. Σαν να ήταν μία τροπολογία ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για να έχουμε το ασφαλέστερο δυνατό αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Περισσεύει όμως ένας από το ΕΛΚ. Ξεκολουθεί να περισσεύει ένας από το ΕΛΚ, ένας παραπάνω. Ο κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ πολύ. Που σημαίνει το αποτέλεσμα, το τελικό 30 υπέρ, 50 κατά, 0 αποχές, καμία αποχή. Πάμε τώρα ε, στην τελική ψηφοφορία και ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, Ψηφίζουμε πάλι ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. And the vote, the end vote on the... Λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα, πάλι ένας από το άλλο και περισσεύει παρακαλώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέκερ που αποσύρεστε. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα 28 υπέρ, 20 κατά, και δύο αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ για το αποτέλεσμα. Yes. Ε, thank you for this. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης ε, και ελπίζω να μείνετε στην αίθουσα για να παρακολουθήσετε το επόμενο θέμα. Ένα λεπτό μόνο για να φύγουν όσοι επιθυμούν να φύγουν. Θα περάσουμε στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.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 Thank you. And uh, now we are coming to uh, uh, on the agenda. Um, Πάμε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα παρακαλώ να καθίσετε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στον εισηγητή μας για το θέμα αυτό, για το συντονισμό των συστημάτων ε, κοινωνικής ασφάλισης, τον κύριο Μπάλας. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν μπω στην ουσία της συζήτησης, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμότατα όλους τους κοιόδης συζητητές ε, που ε, κατέθεσαν τροπολογίες αλλά και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 600 τροπολογίες έχουμε πια για την συγκεκριμένη έκθεση που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, καταλαβαίνετε. Ε, εγώ ήμουν και εισηγητής ε, για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ήταν πάνω από 700 τροπολογίες τότε. Οι 600 λοιπόν δεν με φοβίζουν. Ε, είχαμε δουλέψει με την Τανούτα τότε και είχαμε συνεργαστεί πολύ καλά. Έχω διαβάσει το σύνολο των ε, τροπολογιών αυτών και θα ήθελα να σας πω σήμερα ποια ε, είναι η πρώτη σύνοψη που μπορώ να κάνω από ε, τις συζητήσεις που κάναμε για ένα ζήτημα που είναι περίπλοκο γιατί υπάρχουν διάφορα σημεία στην πραγματικότητα τα οποία δεν συνδέονται υποχρεωτικά το ένα με το άλλο. Καταρχάς, να ξεκινήσω ποια ήταν η ιδέα της Επιτροπής ε, κατά την ε, ε, παρουσίαση αυτής της αλλαγής του συστήματος ώστε να εναρμονιστούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δηλαδή όταν κάποιος μετακινείται στην εργασία του να μπορεί να έχει την κοινωνική του ασφάλιση δεν εναρμονίζουμε, συντονίζουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά κοινωνικά συστήματα ανάλογα με τις διάφορες ε, χώρες ε, βέβαια, γιατί δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία, τις οποίες αφορά αυτό το συντονισμό που θα συζητήσουμε σήμερα. σας πω λοιπόν τις πρώτες μου παρατηρήσεις για τις, ε, για τις, ε, πρώτες... για τις πτυχές που θεωρώ ότι είναι σημαντικές για το θέμα αυτό. Καταρχάς, συντονισμό των επιδομάτων ανεργίας. Πρώτον, όσον αφορά την εξαγωγή των επιδομάτων ανεργίας, δηλαδή ένα άτομο άτομο που πηγαίνει στο εξωτερικό να ψάξει μια θέση εργασία μπορεί να έχει δικαίωμα επιδόματο ανεργία κατά τη διαμονή του στο εξωτερικό. Αυτό επεκτείνεται από τρει-έξι μήνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα πρόταση και αφήνει στην, ε, στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα μέχρι την εκπνοή ε, τη ε, περίοδου των δικαιωμάτων. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη πρόταση και προτείνω μάλιστα να επεκτείνουμε αυτή την εξαγωγή μέχρι το τέλο του επιδόματο ανεργία το διαβάσατε αυτό και υποβάλλατε και σχετικές τροπολογίες. Υπάρχουν τροπολογίες ε, που δείχνουν μια τεράστια διάσταση απόψεων ε, ε, μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Κάποιοι, οι, κάποιες υποστηρίζουν την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλες προτιμούν να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, άλλες ομάδες εργασίας θέλουν ε, πλήρη εξαγωγή των δικαιωμάτων. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία, ενδεχομένω να καταλήξουμε με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω, είναι κάτι πρέπει να συζητηθεί μεταξύ μας. Ε, εγώ ε, ξέροντας ε, τις διαστάσεις απόψεων ε, θα έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα μεταξύ των πολιτικών ομάδων και εγώ δεν θα ήθελα να έχουμε φιλοδοξίες πέρα από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για την ε, επέκταση στους έξι μήνες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την μελέτη που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και ε, της Υπηρεσίας Έρευνας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λέει ότι η περίοδος, η μεγαλύτερη επιδομάτων ανεργίας αυξάνει τις πιθανότητες να βρει κάποιος μια θέση εργασίας. Θα ήθελα να το συζητήσω με συναδέλφου ε, που το επιθυμούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά τώρα την άθρηση ή την ομαδοποίηση, ε, η τελευταία δραστηριότητα του ετούντο θέση εργασία πρέπει να δει ε, την τελευταία δραστηριότητά του σε ποια χώρα είχε λάβει χώρα για τουλάχιστον τρει μήνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατάσταση όμω έχει αυτή τη στιγμή είναι κάπου συγκεχημένη ε, για τι αρμόδιες αρχέ των κρατών μελών. Υπάρχει μια ελάχιστη περίοδος για κάθε κράτο μέλο. Για κάποια κράτη είναι μια εβδομάδα, για κάποια άλλα είναι ένα μήνας, για κάποια άλλα είναι τρει μήνες. Η άθρηση λοιπόν είναι μια από τις αρχές ε, της συγκεκριμένη νομοθεσία. Θα προσπαθήσω να μιλάω πιο αργά. Ε, όπως αναφέρθηκε λοιπόν από την μελέτη το, της ε, Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός από τις διευκρινήσεις, υπάρχει, ε, ενέχει και κάποιους περιορισμούς. Γι' αυτό ζήτησα ένας μήνας να είναι η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας πριν από την άθρηση των ε, περιόδων εισφορών στο κράτος μέλος της τελευταίας δραστηριότητας. Και επί του θέματος αυτού υπάρχει η μεγαλύτερη διάσταση απόψεων. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που έχουν σκοπό να καταστήσουν υποχρεωτική την περίοδο άθρησης από την πρώτη ημέρα όπως ε, η τροπολογία 98 και άλλων ε, ε, συναδέλφων του ΕΛΚ, όπως για παράδειγμα η κυρία Στέφενς από το ECR προτιμά την τοποθέτησή της στην τροπολογία 104. Όσον αφορά λοιπόν την εισφορά και την ελάχιστη περίοδο εισφορών, εγώ είδα την τροπολογία 103 του Εμίλιαν Πάβελ που λέει ότι αυτή η περίοδος ασφάλιτης θα έπρεπε να συμπεριλάβει την περίοδο ε, ικανότητα εργασίας λόγω κάποια ασθένεια ή κάποιου ατυχήματο, ε, γιατί ε, ε, υπάρχουν και πολλές άλλες, επειδή όμως υπάρχουν και πολλές άλλες τροπολογίες που συμπληρώνουν αυτή την ιδέα, θα υπάρξει μια συμβιβαστική τροπολογία. Τώρα, για τους μεθοριακούς εργαζομένους που είναι πολύ επίμαχο ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η χώρα τελευταίας απασχόλησης να δίνει το επίδομα ανεργίας αν έχουν ε, για διάστημα 12 μηνών δουλέψει σε αυτή τη χώρα. Με τους ισχύοντες κανόνες το κράτος κατοικίας ε, είναι αυτό που είναι υπεύθυνο ε, αλλά το εισφορές πηγαίνουν στο κράτος εργασίας και φαίνεται λογικό το κράτος μέλος της δραστηριότητας να είναι αυτό που είναι υπεύθυνο για τις εισφορές όμως θα πρέπει να, γίνουν, να υπάρξουν διευκρινήσει για τις προβλεπόμενες διατάξεις ώστε η εξέλιξη προτείνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καταλήξει σε πρακτικές δυσκολίες ε, διοικητικής φύσεως, γλωσσικής ε, ή ε, παροχής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να προβλέψουν συστήματα οικονομικά για να μπορούν να καλύψουν τα τα κενά ε, μεταξύ του επίπεδου εισφορών και των, της, ε, ε, των επιδομάτων, γιατί υπάρχει περίπτωση τα κράτη-μέλη να χάσουν πολλά χρήματα βάσει της πρώτα Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να βρεθούν σε πολύ περίπλοκες καταστάσεις και νομική φύσεως τη στιγμή που θα πρέπει να διαχειριστούν κάτι τέτοιο με τις εθνικέ αρχέ του κράτους ε, στο οποίο ε, εργάστηκε ο εργαζόμενος. Εντάξει, ε, συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να υπάρξουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τους μεθοριακούς εργαζομένους για να μην υπάρξουν κοινωνικές συνθήκες πολύ κακές. Επίσης θα ήθελα να συζητήσω με τους σκιώδεις συζητητές, με τον κύριο Σούλτσε κυρίως, για τη διατήρηση του συστήματος που ισχύει αυτή τη στιγμή με αποζημίωση, με αντιστάθμιση μεταξύ των κρατών μελών αποτελεσματική Ενό συστήματο à la ε, για τον μεθοριακό εργαζόμενο ή ενός συστήματος ε, ε, πρόσβασης στα επιδόματα ανεργία για τους μεθοριακούς εργαζόμενους διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Όλα αυτά είναι προτάσεις που έχω λάβει από τις τροπολογίες. Όσον αφορά τώρα τη μαχροχρόνια περίθαλψη που έχει να κάνει με τις παροχές ασθενείας. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, τις επαγγελματικέ οργανώσεις, τους δικαιούχους, ειδικότερα ως προς την επεξεργασία του καταλόγου των ε, ε, εν λόγω παροχών. Περιμένω να δω κατά πόσο η πλειοψηφία υποστηρίζει ή όχι αυτό το ειδικό κεφάλαιο. απάντηση είναι πάρα πολύ σαφής. Η απαντηση ειναι παρα πολυ σαφή. η τροπολογια 342 από του σκιώδη ηγηγή Σούλτσε ε, από ε, το ΕΛΚ, όπω επίση και από πολλούς ε, ευρωβουλευτές, διαφωνεί. 344 Λάμπερτ επίσης, διαφωνεί. Από την κυρία Χάρτιν επίσης διαφωνεί. 346 της σκιώδης εισηγήτρια και πρόεδρο Γκουε τη κυρία Τζίμερ και άλλων ευρωβουλευτών τη ομάδα, τη επίση ε, διαφωνεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν πολύ λογικά να καταλήξουμε ότι θα υπάρξει μια τεράστια διαφωνία όσον αφορά τη δημιουργία ενός καινούριου ειδικού κεφαλαίου. Συνεπώς θα χρειαστεί να δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε στο υπάρχον κεφάλαιο αυτές τις νέες προτάσεις ε, ε, σε σχέση με την ε, μακροχρόνια περίθαλψη και τις ασθένειες ε, μακράς διαρκείας με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, με έναν τρόπο εύληπτο από τους χρήστες σήμερα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία και να ε, υπάρξει συνένεση των περισσότερων συναδέλφων. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ενσωματώσει την πρόσφατη νομολογία του δικαστηρίου σε σχέση με την πρόσβαση των φορητών, των μετακινούμενων εργαζομένων σε σχέση με τι ε, εισφορέ κοινωνική ασφάλιση. Ε, λαμβάνω γνώση τη νομολογία, αλλά εμεί ω συνομοθέτε δεν πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε στην κωδικοποίηση των αποφέσεων του δικαστηρίου και νομίζω ότι το Συμβούλιο συμφωνεί μαζί μα. Έχω λάβει υπόψη τις διάφορες τροπολογίες διαγραφής, ε, επέκτασης ε, των παροχών ασθενείας και των ε, ασφαλίσεων ασθενείας στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μην μπούμε σε πολλές συζητήσεις πάρα πολύ δύσκολες που θα καταλήξουν στη δική μας ερμηνεία της νομολογίας. Κάνω προτάσεις σχετικά, αλλά πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είναι δυσανάλογη αυτή η συζήτηση για του διάφορου τους που έχουν θέσει κάποιοι, γιατί ούτως ή άλλως η νομολογία ισχύει όσον αφορά την νομοθεσία που ε, ισχύει, την απόσπαση, την πολλαπλή δραστηριότητα, την επαγγελματική κλπ. Ε, ως προς την τυποποίηση των διαδικασιών για, το φορμό, για την έκδοση, το μορφότυπο ε, των εγγράφων της κοινωνικής ασφάλισης για τον καθορισμό ε, των εγγράφων και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδίδονται όταν υπάρχει ας πούμε μια ακρίβεια η οποία τίθεται να από το κράτος μέλος εργασίας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών των αρμοδίων αρχών μέσω του ορισμού ε, μιας ε, περίοδου ε, απόκρισης στο αίτημα συντομότερης. Ε, Πρέπει να υπάρξει δηλαδή μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν πολύ με τις τροπολογίες, ας πούμε 522 και 523 της ΓΟΕ. Αναφέρομαι επίση και στην τροπολογία της κυρίας Αζέα, ε, μια τροπολογία 5 αστέρων για τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών ε, υποστηρίζω την ύπαρξη νέων μηχανισμών, ε, νέων ηλεκτρονικών δικτύων ε, που θα συνδέουν τα κοινωνικά συστήματα όπως γίνεται στο Βέλγιο, την ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής κάρτας με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και σε γενικές γραμμές είναι απαραίτητο να υπάρξει μια, ένας εξυγχρονισμός ψηφιακός. Κύριε Μπάλας, διακόπτη πρόεδρος τρέχετε πάρα πολύ, είναι αδύνατο να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Οι τροπολογίες 460, 461 και 462 τη ΓΟΥΕ και των Σοσιαλδημοκρατικών και του ΕΛΚ πηγαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και, και χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τους ισχύοντες κανόνες για τους ε, αποσπασμένους, ελάχιστη περίοδος υποχρεωτική ε, ε, ε κοινωνικής ασφάλισης του κράτους ε, αποστολής, 558 και 559 Μωρέν Σαρτιέ και άλλων μελών του ΕΛΚ και την 160 της κυρίας Ατζέα πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση για ε, τα ε, έγγραφα που θα μπορεί να παίρνει μαζί του ο εργαζόμενος σε περίπτωση εργασίας σε ένα άλλο κράτος μέλος. Το ζήτημα τώρα του ενεπιδόματων ε, ε, των οικογενειακών σε σχέση με τον τόπο κατοικία των παιδιών. Είναι μια πρόταση κάποιων κρατών μελών. Να επενθυρίσουμε ότι λιγότερο από 1% των οικογενειακών επιδομάτων ε, πληρώνονται προ ε, παιδιά τα οποία ζουν σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό που δουλεύουν οι γονείς του, συνεπώ ο εντοπισμός ε, και η ενημέρωση των ε, επιδομάτων ανάλογα με το πού ζουν οι γονείς, ε, τα παιδιά, συγγνώμη, θα είχε ως αποτέλεσμα ένα σύστημα πολύ περίπλοκο και πολύ δαπανηρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμφωνεί, κάποιοι ημών δεν συμφωνούμε, το σημειώνω. Θα ήθελα όμως να πω ότι εγώ διαφωνώ με αυτήν την συμπερίληψη, γιατί αυτό σημαίνει μια διάκριση μεταξύ των Ευρωπαίων που ζουν στον ίδιο τόπο, ε, και που πρέπει να έχουν ένα διαφορετικό είδος επιδομάτων. Θα είναι πολύ δύσκολο όμω να το διαπιστώσουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμία στατιστική που να δείξει ότι το άχθο αυτό είναι πολύ μεγάλο για, τις, ε, για τα δημόσια οικονομικά των ε, κρατών μελών. Θα είναι πάρα πολύ περίπλοκο και δαπανηρό ένα τέτοιο σύστημα και νομίζω ότι το ποσό θα είναι υψηλότερο από το όφελο που θα προκύψει για τα κράτη-μέλη που θα ήθελαν να υπάρξει αυτή η συμπερίληψη ε, αυτού του παράγοντα. Ε, φυσικά θα το συζητήσουμε αυτό κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των σκιωδών εισηγητών μεταξύ των ε, και μεταξύ των εισηγητών για να δούμε ε, πώς θα κινηθούμε. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού για το συντονισμό ε, σκοπό έχουμε να αποφύγουμε τη γενικευμένη ε, απάτη, ε, τον, τον καλυμμένο προστατευτισμό αλλά και τον κοινωνικό τουρισμό. Θα δοθεί η δυνατότητα να υπάρξει ε, ένα συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης ποιοτικό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση και νομίζω ότι θα έχει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και συγγνώμη που τα είπα τόσο γρήγορα. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Μπάλας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 ε, αυτά που είπε είναι σωστά. Ε, περίπου 700 οι ε, και αν τις δει κανείς υπάρχουν τα πάντα. Εδώ στην Επιτροπή Απασχόληση, σε σκιώδεις ηγητές, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευέλικτοι αν αναζητούμε κάποια λύση. Και αυτό με ανησυχεί γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διχασμός μόνο στις πολιτικές ομάδε, αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ξεκινάω λοιπόν με αυτά τα οποία κατά την αποψή μου είναι τα λιγότερο επίμαχα. Ε, αναφέρομαι στην ε, μακροχρόνια φροντίδα. Ε, πάρα πολλοί συνάδελφοι αναφέρονται ότι είναι υπέρ της ενσωμάτωσης και σε αυτό στο θέμα της υγείας. Κατόπιν θα ήθελα να μιλήσω και για την κωδικοποίηση των αποφάσεων σχετικά με τους ε, οικονομικά ανενεργούς. Εγώ είμαι υπέρ της ε, κωδικοποίησης γιατί σε τελική ανάλυση να μην υιοθετήσουμε την κείμενη νομοθεσία. Υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ισχύουν για μια σειρά παραμφερών υποθέσεων. Κατά την άποψή μου αυτό προσφέρει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Είμαι αισιόδοξο ε, και γι' αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να οργανώσουμε την πλειοψηφία και να βρούμε τον κοινό παρονομαστή. Επόμενο θέμα, αποσπασμένοι εργαζόμενοι σε τομείς κοινωνικού δικαίου. Ό,τι έχει σχέση με την αντιμετώπιση της απάτης, από αυτού νομίζω ότι μπορούμε πολύ σύμφωνα γρήγορα να συμφωνήσουμε. Εγώ είμαι υπέρ μιας πρακτικής λύσης. Οι βραχυπρόθεσμες αποσπάσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι ε, εύκολες, χωρίς γραφειοκρατία. Οι κανονισμοί τις, τους οποίους πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτούς τους βρίσκω ε, εφικτούς και εφαρμόσιμους. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να να εγγυώνται ότι το έντυπο Α1 μπορεί κανεί να το ζητήσει πριν από την βραχυπρόθεσμη απόσπαση. Εγώ είμαι ανοιχτό για μια τέτοια λύση. Και όσον αφορά και την ε, ενσωμάτωση ενό εργαζόμενου σε ένα σύστημα κοινωνική ασφάλιση πριν από την απόσπαση, αυτό το βρίσκω πολύ λογικό, αν και πρέπει να προσέξουμε οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι να μην περιμένουν πάρα πολύ μέχρι να αποσπαστούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ισχύει το σύστημα της χώρας που αποστέλει. Όσον αφορά τις ε, παροχές ε, για τους ε, ανέργους, νομίζω ότι στο θέμα της ενσωμάτωσης υπάρχουν όλες οι εκδοχές, δηλαδή υπάρχουν ρυθμίσεις μια ημέρα σχετικά με το ποιο κράτος θα πρέπει να είναι αρμόδιο. Ε, ο εισηγητή ε, αναφέρθηκε και σε περίοδο ασφάλισης των έξι μηνών που έχει προηγηθεί. Όσοι λοιπόν μιλάνε και αναφέρονται σε προηγούμενη ασφάλιση ε, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι δεν μπορεί κανείς να επιθυμεί μια γενναιόδηρη ε, προασφάλιση ε, και μετά να είναι αρκετά συντηρητικός. Γιατί στην περίπτωση αυτή νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την ενσωμάτωση και τις εξαγωγές. Κατά τα άλλα, πολλοί λένε τι θα κάνουμε με ένα ανεργό ο οποίος σε διάφορα έχει εργαστεί λιγότερο από τρεις μήνες. Δηλαδή ο άνεργος αυτός ε, ε, πώς θα μπορέσει να βρει ένα κράτος μέλος όπου επιτέλους ε, να μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Και το τρίτο που είναι επίσης σημαντικό, διαχωρίζουμε πλέον τις παροχές είδους είδος και τις παροχές σε χρήμα. Αυτό που είπε και ο σχετικά με την ε, αυτο, τη αυτοματοποίηση του επιδόματος ε, τέκνων. Ε, όλοι λένε αυτό θα πρέπει να γίνεται αναπαιδί και εγώ να σας εξηγήσω γιατί όλα αυτά τα βρίσκω σωστά. Πρώτον, και αυτό πρέπει να το πούμε, ο David Cameron δέχθηκε ή απέσπασε την υπόσχεση αυτή από τα άλλα κράτη-μέλη για να παραμείνει η Βρετανική Ένωση στην ε, η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί αυτό ίσχυε παλαιότερα και τώρα δεν ισχύει πια. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους το πώς θα χορηγούνται τα οικογενειακά υποδέματα. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τιμαριθμοποιεί ε, τα επιδόματα, τα κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα τέκνων, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη στο Λουξεμβούργο. Και αυτό θα πρέπει πάλι να το εξηγήσουμε στου ε, πολιτέ, γιατί για κάποιου ισχύει και για άλλου όχι. Κατά τα άλλα, ε, τα υψηλά επιδόματα τέκνων, ε, αυτά δάσονται σε κάποιο βαθμό στους ε, μισθούς. Ε, κατά την άποψή μου όμως αυτό είναι κοινωνικό dumping και αυτό το αναφέρουν αρκετά κράτη-μέλη που ε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και πέμπτον, οι χώρες που είναι κατά της τιμαριθμοποίησης, αυτοί το κάνουν ήδη σήμερα και θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα, πρέπει να συζητηθούν. Υπάρχει λοιπόν μία ομάδα κρατών που έχουν ανώτατο όριο εισοδήματο ως κριτήριο για την καταβολή επιδόματος τέκνων και άλλων οικογενειακών επιδομάτων. Δηλαδή αν ο ένας γονέας είναι πάνω από αυτό το όριο στην ε, χώρα του προέλευση, δεν παίρνει τίποτα. Αν ο άλλος γονέας ζει ε, στο εξωτερικό πρέπει να ε, βάζει το σύνολο του επιδόματος ε, και όχι τη διαφορά όπως, ε, είναι το, όπως προβλέπει το κείμενο ενωσιακό δίκαιο. Αυτό είναι πρόβλημα κατά την άποψή μου. Ορισμένα κράτη-μέλη χορηγούν διευκολύνσεις στο βαθμό που ε, το παιδί ζει με τους ε, γονείς εκεί όπου υποβάλλουν ε, την φορολογική τους δήλωση. Άρα δηλαδή το παιδί θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια χώρα με τους γονείς. Αυτό κατά την άποψή μου περιορίζει την κινητικότητα γιατί στην περίπτωση αυτή οι γονείς θα σκεφτούν και άλλη μια φορά το κατά πόσο θα καταλήψουν τη δουλειά τους για να πάνε σε άλλη χώρα. Και ένα τρίτο θέμα. Υπάρχει ένα κράτος μέλος το οποίο δεν καταβάλει επίδομα τέκνων στην επικράτειά του αν οι γονείς παίρνουν επίδομα τέκνων από το εξωτερικό. Αυτό είναι έμεση διακριτική μεταχείριση και πρέπει να το εξετάσουμε. Και τελευταίο σημαντικό θέμα επ' αυτού υπάρχει ένα κράτος μέλος ε, το οποίο ε, φορολογεί επιδόματα που παίρνουν οι γονείς από άλλα κράτη-μέλη. Τα επιδόματα όμως που έρχονται από το εξωτερικό κατ' ουσίαν έχουν το στόχο να στηρίξουν τα παιδιά ε, και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως φορολογήσιμο εισόδημα γιατί αυτό είναι παράνομο και αυτά τα θέματα ζητάνε όλοι τον ομιλητή να μιλήσει πιο αργά ο ομιλητής δυστυχώς συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό πάμε πάρα πολύ το θέμα λοιπόν δεν είναι να υπάρχει διακριτική μεταχείριση και όσον αφορά το 1% νομίζω το γνωρίζουμε εντωμεταξύ ότι η φορολογητέα βάση κατά την άποψή μου δεν είναι σωστή. Εκείνο που έχει σημασία είναι με το θέμα αυτό να ασχοληθούμε, να βρούμε κάποια λύση και τα θέματα τα οποία σας παρουσίασα αυτά να μην τα αγνοήσουμε. Νομίζω ότι πριν από λίγο καιρό το ανακοίνωσα αυτό και στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πριν περάσουμε στην κυρία Στίβενς, ε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάτε λίγο πιο αργά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους διερμηνείς. να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν. Κυρία Στίβενς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ θα μιλήσω αργά για να μπορέσω να μιλήσω στα Ολλανδικά και να με καταλάβουν όλοι χωρίς κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για, για, στο ότι έχουμε να κάνουμε μια σημαντική μεταρρύθμιση του, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ως προς το συντονισμό τους έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και μια πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρώπη είναι και δίκαιη και κοινωνική και επίσης ε, η εσωτερική ε, αγορά ε, μπορεί να φέρνει κάποια πλεονεκτήματα αλλά αυτό δεν σημαίνει κατάχρηση της κοινωνικής ασφάλισης ούτε κοινωνικό τουρισμό ε, πρέπει να στείλουμε λοιπόν αυτό το πάρα πολύ ηχηρό μήνυμα προ όλου. Γι' αυτό ακριβώ υποστηρίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αποσκοπεί τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να εγγυηθούν την πρόσβαση στι κοινωνικέ παροχέ ε, αλλά να υπάρχει ένας ε, ε, να υπάρχει ειδική ρύθμιση για τους μετακινούμενους εργαζομένους. Ε, πρέπει πρώτα λοιπόν να υπάρχει μία εισφορά σε ένα κοινωνικό σύστημα πριν μπορέσει να έχει επιδόματα, ε, να λάβει επιδόματα, γιατί διαφορετικά το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μακροχρόνια δεν θα μπορέσει να ε, να ε, επιβιώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο και την, κυκλοφορία, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως αυτό να γίνει με κάποια όρια. Θέλουμε να στοχεύσουμε ειδικότερα αυτό τον τουρισμό των κοινωνικών παροχών. Δεν θέλουμε να ε, καταργήσουμε δικαιώματα για τους πολίτες μας. Γι' αυτό ακριβώς υποστηρίζω την ιδέα του να υπάρχει μία μικρή περίοδος ε, τριών ή έξι μηνών, δεν έχει πολύ σημασία, αλλά μία περίοδος αναμονής πριν ένας εργαζόμενος ε, μετακινούμενος να μπορέσει να ζητήσει ένα επίδομα στο κράτος μέλος που τον υποδέχεται. Όσον αφορά αυτή τη φορητότητα των ε, επιδομάτων ανεργίας, εγώ δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμη η επέκταση σε έξι μήνες. Αντιθέτως θεωρώ ότι δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες όσον αφορά τον έλεγχο ο πολίτης που θέλει να μετακινηθεί και που λέει ότι πρέπει να έχει φορητότητα στα δικαιώματά του ε, έχει πλέον και κάποιες τεχνολογικές δυνατότητες ε, να ζητήσει μία θέση εργασίας σε ένα άλλο κράτος μέλος χωρίς να μεταβεί όντω ε, στο άλλο κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το ζήτημα της ε, τιμαριθμικής προσαρμογής των οικογενειακών επιδεμάτων για τα οποία μίλησε ο εισηγητής, αλλά και άλλοι συνάδελφοι. Να σας πω πώς το βλέπω εγώ. Σας το λέω ειλικρινά. Εγώ συμφωνώ με τέτοιου είδους τιμαριθμική προσαρμογή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό το παιδί να έχει τα δικαιώματά του, να έχει την ίδια υποστήριξη για την εκπαίδευσή του και τη συντήρησή του. Ε, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίζεται τον ίσο μισθό για ίση εργασία στο ίδιο επίπεδο, αλλά δεν υπερασπίζεται το δικαίωμα της, του ίδιου επιδόματος για το κάθε παιδί όπου και αν βρίσκεται. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση κατά τη γνώμη μου. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και στο θέμα της απόσπασης. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο εξής ότι οι απάτες είναι βεβαίως απαράδεκτες και πραγματικά θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου ε, το δικαστήριο είπε ότι ο εθνικός δικαστής δεν μπορεί να δεχθεί το έγγραφο Α, ας πούμε, αν είναι αντικείμενο μίας απάτης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, στην οποία πρέπει να στοχεύουμε και συνεπώ είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι η αρχή αυτή που προκύπτει από την ομολογία να θεσμοθετείται και μέσω τη νομοθεσία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό το θέμα, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όμω είμαι πεπισμένη ότι όλοι μας έχουμε συμφέρον να καταλήξουμε σε ένα εξισορροπημένο κείμενο και θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω επικοδομητικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Στέβενς. Κυρία Χάρκιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ σφαιρική εικόνα που μας δίνει με την πρόταση και με τις τροπολογίες. Ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης στόχο έχει για μένα πάνω απ' όλα ένας πολίτης ο οποίος μετακινείται από τη μια χώρα στην άλλη για να βρει μια θέση εργασίας να μην κινδυνεύει να ε, μείνει ακάλυπτος γιατί έχει περάσει από το ένα σύστημα στο άλλο και έχει πέσει κάπου στο κενό μεταξύ των δύο. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε να κάνουμε με την λεγόμενη εξαγωγή. Υπάρχουν μια σειρά μελετών που δείχνουν ότι η επέκταση της περίοδου εξαγωγής προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες για εξασφάλιση θέσης εργασίας, για ανέβρεστες εργασίας. Τώρα αν είμαστε ικανοποιημένοι για την πρόταση της Επιτροπής, με την πρόταση της Επιτροπής, ίσως θα ήταν καλό βέβαια να γίνει ε, να βελτιωθεί η πρόταση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δύσκολα μπορούν να παρακολουθήσουν τη δουλειά που την απασχόληση κάποιου στο εξωτερικό. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε δυσκολίες ως προς την ισότιμη μεταχείριση στη χώρα προελεύσεως. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση για την συσσόρευση. Η έχω να πω ότι είμαι ικανοποιημένη από την πρόταση Επιτροπής. Θα πρέπει βεβαίως να εξασφαλιστεί η προστασία των ε, διασυνοριακών εργαζομένων και στο τελικό κείμενο να μην προκύπτουν από το τελικό κείμενο να μην προκύπτουν ε, δυσκολίες διοικητικές περιτές. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι ανησυχώ πως μπορεί να είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα για τους διασυνοριακούς εργαζομένους μπορεί να μην καταφέρουν τελικά να ε, έχουν κάλυψη των ε, δικαιωμάτων τους και μακροπρόθεσμα. Εμείς δεν υποστηρίζουμε την ε, εγκαθίδρυση ενός ειδικού κεφαλαίου για τη μακροπρόθεσμη προστασία. Είμαστε εν γέννη υπέρ της κωδικοποίησης μέσα και από την ομολογία αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν όλες οι πλευρές. Γιατί μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και εύστοχες όλες οι απόψεις και γι' αυτό θα ήθελα να τις ακούσουμε πριν προχωρήσουμε σε κάποια κωδικοποίηση. Για τους αποσπασμένους, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε πρόταση θα είναι ως το δυνατόν πιο συσταλτική, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ε, της απάτης και απέναντι σε αυτό θα πρέπει να προστατευθούμε για τα οικογενειακά ευεργετήματα. Βεβαίως και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, ανάγκη για την εγκαθίδρυση ενός ε, ε, μηχανισμού επικουρικού σε περίπτωση που αλλού μένουν οι γονείς και αλλού τα κράτη-μέλη για τα οικογενειακά ευεργετήματα. Ο κύριος Σόλτς είπε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε καλά συστήματα που θα λειτουργούν ικανοποιητικά σε διαφορετικά κράτη-μέλη αυτό που θα πρέπει να κάνουμε βεβαίως είναι να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα και να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε μία ε, λύση ή φόρμουλα μία λύση που θα μας ε, επιτρέψει να δώσουμε απάντηση στους προβληματισμούς και βεβαίως περιμένω να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ τον εισηγητή και αναμένω πολλές ε, μακροσκελείς συζητήσεις και συνεδριάσεις. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Λόπες Βερμέιο. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την Γκάμπι Τσίμερ η οποία δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Ε, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις, είναι και πρόεδρος της ομάδας μας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μεταφέρω το μήνυμά της σε γενικές γραμμές υποστηρίζουμε τη θέση του κειμένου του εισηγητή και υποστηρίζουμε την εξαιρετική του δουλειά. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες που σκοπό έχουν να βελτιώσουν επί πολλών σημείων ε, το κείμενο. Τέσσερις αρχές είναι ο γνωμονάς μας για τις τροπολογίες αυτές. Πρώτον, ε, συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων ασφάλισης. Θεωρούμε ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει να διατηρούν όσο το δυνατόν καλύτερο, καλύτερα τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των αποσπασμένων και μετακινουμένων εργαζομένων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, οι κανόνες πρέπει να είναι απλοί, εύληπτοι και για τους πολίτες και για τις ε, αρχές. Να μην υπάρχει δηλαδή πρόσκομα διοικητικό το οποίο θα εμποδίζει του παλο... Ε, τους πολίτες γιατί θα έχουν να αντιμετωπίσουν ε, πάρα πολύ περίπλοκους κανόνες. Τρίτον, δεν πρέπει οι πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωσης να είναι ε, εξορισμού ε, αν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα μετακίνησής τους. Και επίσης πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν, θα είναι θύματα ε, των ε, καταχρήσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων τους από τις επιχειρήσεις. Δεν θα πω σε όλες τις λεπτομέρειες, ε, αλλά θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Πρώτον, όσον αφορά τους ανέργους που αναζητούν ε, απασχόληση, η μη ενεργοί σε, οικονομικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια κοινωνική βοήθεια ή ένα ελάχιστο εισόδημα στο πλαίσιο του κανόνα του συντονισμού, ένα καθεστώς κοινωνικού ε, συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα στους μετακινούμενους εργαζόμενους να υποστηρίζονται οικονομικά. Η ιδέα είναι να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα, ε, τα δικαιώματα των πολιτών μας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ενός εργαζομένου που βρίσκεται σε μια προσωρινή κατάσταση αδράνειας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ε, περιπλέξουμε την πρόσβαση ε, από πλευράς πολιτών. Θέλουμε απλώς να εξαλείψουμε τις διαφορές που υπάρχουν σε διασυνοριακό επίπεδο και μιλάω για την πρόσβαση των διαφόρων, στις διάφορες παροχές στην περίθαλψη κλπ. Όσον αφορά τώρα την κάλυψη για τη μακροχρόνια περίθαλψη, ακούσαμε τα επιχειρήματα εκατέρωθεν ε, και ακούσαμε τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη, υπάρχουν και επίσης και ιδιωτική, υπάρχει ιδιωτική φροντίδα μας λένε ότι το να υπάρξει ένα κεφάλαιο που θα φορά ειδικότερα αυτή την μακροχρόνια περίθαλψη ε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες αστάθμητες, απρόβλεπτες γιατί ε, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην κανονική περίθαλψη με, μια, με έναν ιδιαίτερο ορισμό ε, με συγκεκριμένη διευκρίνηση για το είδος των παροχών που προβλέπονται και αφορά την κάλυψη, την νοσοκομιακή, ε, τις διάφορες παροχές σε περίπτωση διασυνοριακής εργασίας κλπ. Ε, τώρα, η περίοδος των 12 μηνών ε, προτού μπορέσει ο μετακινούμενος εργαζόμενος να ε, θεμελιώσει κάποιο δικαίωμα στο κράτος μέλος εργασίας. Αυτό όμως μπορεί να είναι προβληματικό γιατί μπορεί κάποιος άνεργος να χάσει κάποια δικαιώματά του και το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας. Τώρα, ποιο κράτος μέλος θα δίνει το επίδομα ε, το να το ορίσουμε αυτό θα μείωνε το διοικητικό φόρτο και θα έδινε τη δυνατότητα στους ε, ανέργους να, ε, να βρουν μία δουλειά συντομότερα επίσης. Οι παροχές ανεργίας πρέπει να μπορούν να εξάγονται μέχρι την εκπνοή του επιδόματος ανεργίας για να μπορεί ο εργαζόμενος να έχει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του να βρει μια θέση εργασίας και νομίζω ότι έτσι θα μειώνονταν και πολλά προβλήματα στους μεθοριακούς εργαζομένους. Η εισαγωγή περι... μιας περίοδου τριών μηνών ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το επίδομα ανεργίας πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση και για τις διοικητικές αρχές και για τους πολίτες. Εσείς μιλάτε για ένα μήνα κύριε Σιγητά. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ενδεχομένω ακόμη πιο περίπλοκο και πιστεύουμε ότι για να απλοποιηθεί η ε, κατάσταση κατάσταση. Το άρθρο 101 για το Lex Specialis, για την περίοδο σόρευσης, θα μπορούσε να καταργηθεί και σε σχέση με τις παροχές θα έπρεπε να μιλούμε για το άρθρο 6. Όσον αφορά τα οικογενειακά επιδόματα, πιστεύουμε ότι πρέπει να πλησιάσουμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με, τις, με τα επιδόματα στην περίπτωση για παράδειγμα γονικής άδειας του, της μητέρας ή του πατέρα. Η τροπολογία που έχουμε εμείς καταθέσει αποσκοπεί στη διατήρηση της κατάστασης ακόμη και αν υπάρχει ένας μεθοριακός χαρακτήρας. Ε, είναι επίσης απαραίτητο ο εργαζόμενος να μην φοβάται να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και τα δικαιώματά του πρέπει να γίνονται σεβαστά και βεβαίως ε, στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας και σε σχέση με την απόσπαση πρέπει να, λαμβάνονται ακόμη περισσότερο υπόψη τα δικαιώματα αυτά. Είναι απαραίτητο αν θέλουμε, απαραίτητο αν θέλουμε να έχουμε μία ε, κοινωνία ε, σωστή. Θα ήθελα να πω επίσης ότι εγώ είμαι στη διάθεση του εισηγητή και των ε, υπολείπων συναδέλφων μπορεί να υπολογίζει στη δική μας υποστήριξη για τη δουλειά που έχει να κάνει ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τζιν Λάμπερτ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχουμε κάπως η δουλίτσα. Από ό,τι βλέπω. Καλό θα ήταν να είχε προτείνει ε, ως αναδιατύπωση τα κείμενα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι με τη μορφή που τα κατέθεσε, έτσι θα κερδίζαμε πολύ χρόνο. Δεν θα χρειαστώ να ψάχνουμε σε τι έχει φέρει κάποιες αλλαγές στο νέο κείμενο κτλ. Εν πάση κάποια άλλη φορά. Από τι παρατηρήσει τώρα του εισηγητή και των λοιπόν συναδέλφων θέλω να πω τα Συμφωνούμε με τις προτάσεις ότι δεν πρέπει να υπάρχει χωριστό κεφάλαιο, αλλά ότι πρέπει να μείνει το κομμάτι στο κύριο σώμα. Ως προς το πώς θα γίνει ε, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να τον σηματώσουμε στο τωρινό κείμενο. για να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ως προς μια αναφορά για τον μη οικονομικά ενεργό που ακούστηκε από κάποιους. Εμεί θεωρούμε ότι δεν είναι η νομολογία αρκετά παγιωμένη σε αυτό, άρα θα προτιμούσαμε να βγει. Και επίσης κάποιοι μπορεί να έχουν και διαφορετική αντίληψη προς το τι σημαίνει αυτό σε έννοια νομική. Επομένως, ε, θα προτιμούσαμε να περιορίσουμε το πεδίο και να βγει το κομμάτι αυτό. Ας μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα πολύ αυτή τη στιγμή. Επίσης, ο εργαζόμενος, ο δια και δεν εννοώ τον παραμεθόριο εργαζόμενο εδώ. Αυτός που δουλεύει πέραν των συνόρων. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους που πάνε από το ένα κράτος στο άλλο για τη δουλειά τους. Πάνε για μια συνεδρία για μια μέρα ή μπορεί να αλλάζουν εργοδότη για ένα διάστημα να επαγονται δηλαδή σε κάποιον άλλον. Αυτό είναι μια υποκατηγορία των αποσπασμένων. Και θέλουμε να διπλωσουμε μια πρόταση για να προσθεθεί το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, η οποία θα ήταν ως εξή. Πρώτον, θα έχουμε για τρεις μήνες ανοιχτή ε, ρύθμιση, δηλαδή θα χρειάζεται για κάθε μέρα αυτών των τριών πρώτων μηνών να γίνεται ενημέρωση, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται το κράτος μέλος της υποδοχής όταν κάποιος ταξιδεύει. Αυτό νομίζω μπορεί να μπει στο σύστημα πληροφοριών της ιστορικής αγοράς, γιατί φαίνεται ότι περισσότερο τραβάει την προσοχή των πολιτών κάτι που έχει να κάνει με την εσωτερική αγορά παρά με τα κοινωνικά συστήματα. Αλλά θα συζητήσουμε και με τους κοιόδες Πώς μπορεί δηλαδή το σύστημα να είναι απλό και για αυτόν ο οποίος δεν είναι αποσπασμένος, αλλά και σε σχέση με την ε, οδηγία για τους αποσπασμένους για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Επίσης, για την υπαγωγή στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ε, στο κράτος εργασίας, εμείς προτείνουμε μία περίοδο δίμηνη για να υπαχθεί κανεί στα σχετικά συστήματα και τα δικαιώματα. Για την ε, κάλυψη των οικογενειών, τα ευεργετήματα τα οικογενειακά, Εμεί επεκτείνουμε λίγο περισσότερο αυτό που το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει αναπροσαρμογή των ευεργετημάτων των οικογενειακών. Αρκετά περίπλοκο είναι το σύστημα. Στη τελευταία ανάλυση έχουν, το σύστημα, έχουν τα ευεργετήματα και το κοινωνικό σύστημα που τα συνοδεύει. Οι εργαζόμενοι. Και ας είμαστε και πιο ανοιχτοί στην ιδέα της αλληλεγγύης, αυτό που έχουν πει συνάδελφοι καμιά φορά ότι είναι η βρετανική ματιά. Εμείς δεν θα το υποστηρίξουμε λοιπόν. Πάντως, αντλούμε από τη συζήτηση για τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων το δίδαγμα το σχετικό με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εδώ λέμε ότι πρέπει να μπορεί ο εργαζόμενος ατομικά να υπάγεται στο σύστημα στη χώρα που εργάζεται αυτό πρέπει να είναι απλό, ειδικά και, και προβλέψιμο και ειδικά όταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να προσφέρει ένα σύστημα δεν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Για την επέκταση πρέπει να κοιτάξουμε βεβαίως μέχρι την εξάτληση των δικαιωμάτων, αλλά θα δούμε την ε, ε, τις διατυπώσεις, τις λεπτομέρειες, στο επίδομα ανεργίας. Βλέπουμε ότι η πρόταση πιο πολλά ερωτηματικά για να παραδίνει λύσεις σε προβλήματα. Τροπολογίες έχουμε και σε σχέση με τη Διοικητική Επιτροπή και την πρόσβαση που μπορεί να έχει ο πολίτης για να λύσει τα προβλήματα αυτά που φαίνονται δυσθεώρητα και βεβαίως από ε, εκτελεστικές προτείνουμε να πάμε σε κατεξουσιοδότηση πράξεις με διαφύλαξη των προνομίων των κοινοβουλίων. Αυτά εν ολίγης εκφράζονται μέσα από τις τροπολογίες μας και ελπίζουμε μέχρι το τέλος της θητείας να έχει ολοκληρωθεί η πρόταση. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος ε, του EFTD δεν είναι παρούσα. Τι αντικαθιστά κάποιος. Όχι από ό,τι φαίνεται. Σε εκ τούτου περνάμε στην πολιτική ομάδα ENF στον κύριο Μαρτά. Παρακαλώ. Η κυρία Μελά είναι σκιώδη συγχύτρια, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει και στη συγγνώμη. Πολύ ωραία. Πάμε τότε στον ε, κατάλογο των μελών που επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Βίμπα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του, για την εισήγησή του, την παρουσίαση της έκθεσης. Ε, Προφανώς ε, πρόκειται για πολύ σημαντικό νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καταδεικνύει εξάλλου και το πόσο περίπλοκη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, στα κράτη-μέλη. το να υπάρχει κάποια διαφορετικότητα λόγω των διαφορετικών ιδεολογιών. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ε, σε τελική ανάλυση ε, πολλοί θέλουν μεγαλύτερη κοινωνική προστασία, άλλοι πάλι λιγότερη. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ο διαχωρισμός ε, στα κράτη-μέλη. Η προσέγγιση των κρατών μελών μπορεί να οδηγήσει σε άδικα συστήματα, σε διακριτική μεταχείριση. Ε, Βεβαίως ε, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα, στο θέμα ε, των ε, επιδομάτων τέκνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο χρόνια ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε τέτοιου είδους αναθεώρηση και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αυτό δεν αξίζει για πάρα πολλούς λόγους. Παρ' όλα αυτά Υπάρχουν ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για αυτή την έκθεση και οι τροπολογίες αυτές ε, αναφέρονται στην ε, τιμαριθμοποίηση. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα ότι η τιμαριθμοποίηση μπορεί να ισούται με διακριτική μεταχείριση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις σε όσους έχουν καταθέσει τις τροπολογίες. Η όλη ιδέα είναι η εξής, ότι αν το παιδί δεν εγκαταβεί στον ίδιο χώρο, στην ίδια χώρα όπου ζουν και οι γονείς, τότε το παιδί δικαιούται τα επιδόματα στο κράτος το οποίο εγκαταβεί. Δηλαδή, ας, κάνουμε, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Ε, οι πολίτες ε, που ε, ζουν στην Ολλανδία και έχουν ένα παιδί στην Αρούμπα, τότε το παιδί θα παίρνει τα οικογενειακά επιδόματα της Αρούμπα οι σε ζουν στο Μπουρούντι. Τότε τα επιδόματα με βάση τι θα κρίνονται τα επιδόματα του Μπουρούντι. Δηλαδή, θέλω να πω το εξή Αν δεν θεωρεί κανείς ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από ένα άλλο κράτος μέλος ε, ε, αφήνουν το παιδί στη χώρα τους ε, και να ρυθμίζουμε με βάση αυτό, αυτό είναι διακριτική μεταχείριση. Ή αν θέλετε ένας γερμανός εργαζόμενος που εργάζεται στη Ρουμανία, στη χώρα μου, και κερδίζει λίγο παραπάνω από τον μέσο μισθό της ε, Ρουμανίας. Αν το δικό του το παιδί ε, παραμένει όμως στη Γερμανία, πώς λύνεται το πρόβλημα. θα αναγκάσει κανείς τον Ρουμανό εργοδότη, Ρουμάνο με εργοδότη να καταβάλει τα επιδόματα που ισχύουν στη Γερμανία και να πω και κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος ρεαλισμού. Μιλάμε για το 1% των παιδιών που ενδεχομένως να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να δαπανάμε τόσα πολλά χρήματα για να συστήσουμε έναν τόσο περίπλοκο μηχανισμό ή μήπως ε, επειδή έρχονται οι εκλογές ε, θέλουμε να δώσουμε κάτι, να προσφέρουμε κάτι σε κάποιους πολίτες, σε κάποιες χώρες. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στις αρχικές μας απόψεις του τι είναι δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λένες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για ένα από τα θέματα της νομοθεσίας για τους μεθοριακούς εργαζομένους είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι σημαντική νομοθεσία γιατί έχουμε εδώ τη δυνατότητα για τους ανθρώπους που δουλεύουν σε μεθοριακές περιοχές ε, ε, να μπορούν να δουλεύουν ε, με μεγαλύτερη ευκολία και στην άλλη πλευρά των συνόρων ε, θα πιστεύω ότι πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αυτήν την ε, ευκαιρία. Έχουμε κάνει λοιπόν την εξή επιλογή μέσω των τροπολογιών μας. Όταν κάποιο για πέντε χρόνια δουλεύει σε ένα κράτος μέλος ε, και μπαίνει στην ανεργία, να μπορεί να διαλέξει σε ποιο κράτος μέλος θα λάβει το επίδομά του και αυτό δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθεί ένας δεσμός με την αγορά εργασίας όπου υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για αυτόν να βρει μια δουλειά. Δυστυχώ, αυτό δεν είναι πάντοτε πολύ εύκολο για τους ε, μεθοριακού εργαζομένους. Πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Είναι περίπλοκες οι συνθήκες για αυτού τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει μια ε, λύση προσαρμοσμένη στη δική τους κατάσταση. Γιατί αυτό που είναι τέλειο για τον έναν μπορεί να είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον άλλον. Επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε όλες τις επιλογές και η επιλογή αυτή θα ήταν η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων και οι καλύτερες, οι περισσότερες ευκαιρίες έβρεσης εργασίας προκειμένου να ενισχύσουμε τη μεθοριακή, την εργασία ε, στις, παραμεθόριες, στις μεθοριακές ζώνες. Ε, πρόκειται λοιπόν για δικαιώματα ε, περίπου 800.000 ατόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη και νομίζω ότι στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής της νομοθεσίας θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε και με τη δική τους ε, τύχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τη δουλειά του. κυρίως όμως ε, να τους ευχαριστήσω για τη δουλειά που μένει ακόμη να γίνει. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στο κεφάλαιο που αφορά τις συνθήκες πρόσβασης ε, στις παροχές ανεργίας για ε, τους μετακινούμενους εργαζομένους και πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής πηγαίνει σε γενικέ γραμμές ε, προς την ε, σωστή κατεύθυνση και όταν μιλάμε για την επέκταση σε έξι μήνες της, δυνα... των... Ε, δυνατότητας αυτών των δικαιωμάτων σε επίδομα ανεργία, να επικροτήσω επίσης την ελάχιστη περίοδο δραστηριότητας τριών μηνών στη χώρα προέλευση για να μπορεί κανεί να έχει πρόσβαση στο επίδομα ανεργία. Θα ήθελα όμω όμως κυρίως να επιμείνω, όπως είπε και ο συνάδελφος Λέρενς, Λένερς για την κατάσταση των μεθοριακών εργαζομένων ε, είναι πολύ ε, στην Ανατολική Γαλλία που είναι η δική μου εκλογική περιφέρεια. Θα ήθελα να τονίσω και να πω ότι συμφωνώ με την περίοδο μιας ελάχιστης δραστηριότητας 12 ε, μηνών ώστε να γίνει, πριν να γίνει μία μεταφορά ε, σε μία άλλη χώρα του δικαιώματος ε, ε, επιδόματος ανεργίας. Γιατί αν η κατάσταση, η γεωγραφική τους κατάσταση οδηγεί τους μεθοριακούς εργαζομένους προς τη γειτονική χώρα, ακόμη και αν είναι πολύ δραστήριοι και μετακινούνται συνεχώς, νομίζω ότι το μεγαλύτερο συμφέρον τους βρίσκεται στην χώρα κατοικίας. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε αυτήν την ευκαιρία να διαλέξουν, να εγγραφούν στην υπηρεσία ευρέσεως εργασίας της χώρας κατοικίας τους ή διασυνοριακή ε, υπηρεσία έβρεσης εργασίας ε, που υπάρχουν ε, στα σύνορα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι μεθοριακοί εργαζόμενοι, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κατάρτιση, να συμμετέχουν σε επαγγελματική κατάρτιση, να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη γλώσσα τους και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουμε ε, με στόχο βεβαίως ε, την επιστροφή τους ε, στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ντέτσε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γκίον Μπαλά για την έκθεση είναι πολύ καλή. Η αναθεώρηση των εθνικών ασφαλιστικών, κοινωνικών ασφαλιστικών συστημάτων είναι μαζί με την οδηγία για την απόσπαση ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουμε να πραγματευτούμε στην τρέχουσα θητεία. Θα ωφελήσει βέβαια ε, η πρόταση την ε, δυνατότητα κινητικότητα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και βέβαια υπάρχει μια σειρά από ε, ζητήματα που θα πρέπει να απαντηθούν και για τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και για τα κράτη-μέλη. Ισομερή σε παραδείγματι κατανομή της επιβάρυνσης για τα κράτη-μέλη είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης η δυνατότητα υλοποίησης των διατάξεων σε κάθε τομέα και όλα τα κράτη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω ρητά να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαλά για την πρόταση για εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ευρωπαϊκού Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να υπάρχει δυνατότητα του ελέγχου της, ε, εργασιακής σχέσης, του, των συνθήκων εργασίας και βέβαια για να υπάρχει παρακολούθηση του πόσο επιβαρύνονται τα εθνικά ασφαλιστικά συστήματα. Ο εξυγχρονισμό των συστημάτων μπορεί να λάβει χώρα στην πραγματικότητα μόνο εάν οργανωθεί κατά τρόπο σωστό και ικανοποιητικό η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Σε σεβασμό βέβαια και των δικαιωμάτων ε, και των δεδομένων των εργαζομένων αλλά και με διαφάνεια. Βεβαίω, χρειάζεται να προχωρήσουμε ταχύτατα στην ψηφιακή ανταλλαγή δεδομένων για να αποφύγουμε την καταστρατήγηση του δικαίου. Ε, πρέπει να υπάρχουν σαφείς προθεσμίες για την ενημέρωση από το κράτος, υποδοχή στο κράτος ε, προελεύσεως και την υπαγωγή στα δικαιώματα αναλόγως ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπα, πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα. Πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων και να μεριμνήσουμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών. Ε, thank you. Ε, then give the... Ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μπέκερ, ο οποίος επανέλθε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές. Όλος ιδιαίτερος. Είναι πολύ καλή δουλειά για τα κοινωνικά συστήματα. Πολύ επαγγελματική. Βεβαίως και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Σούλτσε, τον ε, σκιώδη συγκητή από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο οποίο με τη δουλειά του συνδυάζει όλε τις προτάσει μα. Εδώ τι έχουμε να παρατηρήσουμε, πρόκειται για έναν τομέα που έχει να κάνει με την αναπροσαρμογή των οικογενειακών δικαιωμάτων, ε, επιδομάτων. Δηλαδή εκεί όπου κανείς έχει να καταβάλει τα έξοδα, τις δαπάνες Διαβίωση των τέκνων του. Περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά. Εκεί πρέπει να έχουμε το κριτήριο που πληρώνει κανείς για να ζουν τα παιδιά του και αναλόγως ε, με το κράτος αυτό θα πρέπει να γίνεται και υπολογισμό των επιδομάτων. Βεβαίω ξέρουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Ασφαλώς πρέπει να ε, εξετάσουμε την υπόθεση, πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε δηλαδή ένα νομικό πλαίσιο για την ε, προσαρμογή και τον υπολογισμό των οικογενειακών επιδομάτων ε, σε σχέση με την αυστριακή πρόταση. Θέλω να επισημάνω ότι δεν κατατίθεται πρόταση για δεσμευτική, δηλαδή υποχρεωτική για όλα τα κράτη ρύθμιση της, αναπροσαρμογής των, της προσαρμογής των ε, επιδομάτων, αλλά αφήνει στο κάθε κράτος την επιλογή της ε, ε, εγγραφής, της προσυπογραφής στο σύστημα. Ο καγκελάριος μου δηλαδή, Σεμπάστιαν Κούρτς, μπορεί να ε, προτιμήσει να πει ότι όσοι μένουν στην Αυστρία παίρνουν αντίστοιχα και προερχόμενοι από άλλα κράτη, παίρνουν αντίστοιχα τα οικογενικά επιδότηματα, αλλά αυτό, επιδόματα, αλλά αυτό θα ισχύει για την Αυστρία μόνο. Πάντως, Θέλω να πω ότι αυτές οι επιλογές θα πρέπει να είναι αμφίδρομες, δηλαδή κάποιο κράτος μπορεί να χρειαστεί να καταβάλει περισσότερα επιδόματα σε κάποιον που ε, προερχόμενος από φθηνότερο κράτος μένει σε αυτό ή το αντίστροφο. δεν πρέπει να επιτρέψουμε τις διαστρεβλώσεις, τις τρεβλώσεις της κατάστασης. Για, το, για την Αυστρία πρόκειται για 250, για 250 εκατομμύρια ευρώ για να μην πω 300 του 2016 με βάση τα στοιχεία που έχω. Και άρα μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια επιλογή θα οδηγούσε σε μείωση του ποσού αυτού στο μισό του, εάν δεν χρειαζόταν να κάνουμε εμβάσματα σε άλλες χώρες για παιδιά που μένουν εκεί ενώ οι γονείς τους εργάζονται στην Αυστρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μένα θα έπρεπε εδώ και καιρό, θα όφιλε εδώ και καιρό να έχει κάνει προτάσεις που θα εξασφάλιζαν ασφάλεια και σαφήνεια του δικαίου. Δεν το έχει πράξει και σε αυτό νομίζω στηρίζεται και η σχετική προφορική ερώτηση των συναδέλφων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλιστεί ακριβώς σαφήνεια και διαφάνεια. Ε, πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να έχουμε μια σαφή δίκαιη και αποδεκτή για κάθε πλευρά ε, πρόταση με βασισμένη πάνω σε θεμητά επιχειρήματα βεβαίως και ελπίζω οι συνάδελφοι να την υποστηρίξουν. Ο κύριος Γκέρικε, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και για την εκτενέστατη έκθεση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να συγκρίνουμε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως όταν πρόκειται για οικογενειακά επιδόματα ε, θα πρέπει να υπάρχει και κάποια εξισορρόπηση ανάμεσα σε αυτούς που δεν έχουν παιδιά και σε αυτούς που έχουν παιδιά. Εδώ πρόκειται για το επίδομα τέκνων. Για σκεφτείτε 5,9 ε, δις ε, οικογενειακά επιδόματα στο εξωτερικό χορηγούνται από μια χώρα το 1,5 είναι επίδομα τέκνων. Αυτό είναι περίεργο, αλλά έτσι είναι. Η Γερμανία το κάνει αυτό και με βάση τις ενωσιακές διατάξεις, διατάξεις που συζητάμε εμείς σήμερα. Περίπου 200.000 παιδιά στο εξωτερικό παίρνουν επίδομα από τη Γερμανία και ε, ε, συνήθως αυτά βρίσκονται στην Πολωνία, Τσεχία, Κροατία. Εκεί βρίσκονται τα παιδιά κατά κανόνα. Για τις οικογένειες σημαίνει για το πρώτο και δεύτερο παιδί κάθε μήνα 94 ευρώ, για το τρίτο 198 και για το περαιτέρω παιδιά περίπου 320 ευρώ. Και να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή 641 ευρώ είναι στη Ρουμανία ο μέσος μισθός. Άρα δηλαδή σας αναφέρω αυτά τα στοιχεία για να σας δείξω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο εντοπίσαμε εμείς και πρέπει να συζητήσουμε κατά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης στην Ευρώπη. Και βεβαίως θα δώσω δίκιο στους συναδέλφους από το ΕΛΚ. Στην Ευρώπη θα πρέπει να μπορούμε να διερωτηθούμε κατά πόσον μια χώρα, ένα κοινωνικό επίδομα ε, θα πρέπει να το καταβάλει σε ένα παιδί τη στιγμή που το παιδί δεν ζει πια στη χώρα ή που ε, επειδή είναι παιδί αλλοδαπών ή γονέων που ζουν στο εξωτερικό δεν έχει ποτέ σε αυτή τη χώρα προέλευσης. Ε, μήπως θα ήταν πιο δίκαιο να υπάρχει τουλάχιστον μία αναπροσαρμογή και η ε, τα επιδόματα να προσαρμόζονται στο κόστος διαβίωσης μια χώρα, αλλά και σε άλλα στοιχεία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε αυτά τα στοιχεία υπόψη μας, να συζητήσουμε για αυτό το ερώτημα, γιατί είναι τα ερωτήματα που τίθενται για τους ε, πολίτες μας και σε τελική ανάλυση εγώ εξελέγω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκπροσωπώ αυτούς τους πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να πω ότι καθόλου δεν ζηλεύω τον εισηγητή μας. Γιατί πραγματικά δεν είναι εύκολο αυτό που έχει να κάνει. Πολύ διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Όμως, είμαστε εδώ ως ε, ε, εκπρόσωποι των πολιτών μας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είμαστε εθνικοί βουλευτές, είμαστε εδώ για να συντονίσουμε ε, τα πράγματα. Ο κύριος Γκέρικε μίλησε για την οικογένεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχετικά επιδόματα, όχι μόνο για την κατάσταση στη Γερμανία. Αυτό είναι σημαντικό. γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ε, να ξεφύγουμε λίγα και αν πάρουμε ως ε, ε, σημείο αναφορά στην κατάσταση σε μία χώρα μόνο. Έχουμε κάποιες υποχρεώσεις και δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις όταν έρχονται εργαζόμενοι σε εμά, στη δική μας χώρα, τους χρειαζόμαστε, πληρώνουν φόρους και έχουν και δικαίωμα σε παροχές. Είναι πολύ λογικό. Πληρώνουν φόρους, όπως ακριβώς και οι ε, πολίτες ε, της χώρας. Υπάρχουν βέβαια κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα για κάθε χώρα και πρέπει φυσικά να βρεθεί μια ισορροπία. Δύο σημεία. Δύο απόψεις μάλλον. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι τα οικονομικά, τα οικονομικά επιδόματα πρέπει να είναι αντικείμενο τη αριθμική προσαρμογή, αλλά υπάρχουν και άλλα επιδόματα που να μπορούμε να τα μετεχειριστούμε με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, τα συντοξιδιωτικά δικαιώματα. Ε, τι θα κάνουμε με αυτά. Τι θα κάνουμε. Ε, θα τα αποκλείσουμε και αυτά. Και με τα επιδόματα ενεργείας θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο, να τα βάλουμε κατά μέρο και να έχουμε ειδικέ ρυθμίσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι είμαστε υπεύθυνοι και σε σχέση με τις παροχές αυτές. Γιατί έχουμε δανούς που θα πάνε στην Ισπανία για παράδειγμα για ένα μήνα για έξι μήνες, συγγνώμη, ε, με τις παροχές τους πλήρως καλυμμένες, γιατί πρέπει να καταγραφούν στο σύστημα της Ισπανίας. Λοιπόν, οι αρχές, η αρχή αυτή περί τριών μηνών είναι μεν σημαντική, αλλά πρέπει να συνεισφέρει κανείς και στη χώρα. Να μην φτάσουμε λοιπόν σε μια κατάσταση αντίστροφη τελικά. Πιστεύω ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι κάτι το δίκαιο και το λογικό. Αυτό θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Να αποφύγουμε κάθε είδους διάκριση. Βάσει της εθνικότητας. Ευχαριστώ πολύ ο κύριο Σούλτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, να απαντήσω γιατί δύο συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε μένα. Ξεκινάω με εσά. Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα επίδομα σε μια παροχή υπηρεσία για, για σύνταξη, δηλαδή και εγώ καταβάλω κάτι και μετά έχω κάποια δικαιώματα. Ενώ όσον αφορά το οικογενειακό επίδομα, ε, σε πάρα πολλέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτω αδιάφορο αν κερδίζω 1.000, 3.000 ή 5.000 ευρώ. Ε, θα παίρνω το ίδιο οικογενειακό επίδομα, γιατί είναι μια παροχή για την οποία δεν έχω καταβάλει χρήματα. Είναι επιπρόσθετο κοινωνικό επίδομα. Ε, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν θα έλεγα ποτέ να αναπροσαρμόζουμε συντάξει για μια παροχή δηλαδή για την οποία έχω καταβάλει εισφορές. Και κυρία Πρόεδρε, αναφέρατε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω αναφερθήκατε στο Μπουρούντι ή σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σε αυτές τις χώρες όλα τα κράτη-μέλη με αυτές τις χώρες έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις. Η Γερμανία, ας πούμε, έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις με πολλές χώρες και εκεί αναφέρεται η αναπροσαρμογή ή και τίποτα. Ή και ούτε καν ε, επίδομα τέκνων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 28 χώρες με 28 διαφορετικές νομοθεσίες ε, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τους πολίτες μας. Αυτό που είπατε εσείς ε, είναι συνάρτηση της συμφωνίας που έχει κάνει μία χώρα χώρα ε, με την τρίτη αυτή χώρα. Και να πω και κάτι άλλο που αφορά στο σύστημα του να εργάζομαι σε άλλη χώρα από αυτήν που παίρνω το κοινωνικό ε, επίδομα. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε καμία χώρα, δεν θέλησα να ονοματίσω καμία για ευνόητους λόγους. Ε, λοιπόν, ζείτε σε μία χώρα με το παιδί σας και έχετε δικαίωμα σε 100 ευρώ επίδομα τέκνου και ο σύντροφος ζει σε άλλη χώρα ή η σύντροφος στη Γερμανία δικαιούται κανείς επίδομα 190 ευρώ. Σε κανονική περίπτωση τα 100 ευρώ τα παίρνετε από τη δική σας χώρα και τη διαφορά αν ζείτε στη Γερμανία θα τα πάρετε από τη Γερμανία. Δηλαδή συνολικά θα πάρετε τα 190 ευρώ ως επίδομα τέκνου. 100 από τη χώρα σας και 90 από τη Γερμανία. Υπάρχει όμως μια κατάσταση όπου ορισμένε χώρες λένε ας πούμε από τα 1000 ευρώ εισόδημα δεν καταβάλλεται πλέον επίδομα τέκνου στην ε, χώρα μου. Και ο εισύντροφος ζει στη Γερμανία τότε ο άνθρωπος αυτός παίρνει παρόλα αυτά τα 190 ευρώ και αυτό είναι διακριτική μεταχείριση κατά των ε, συμπατριωτών γιατί στην περίπτωση αυτή αν έμενε ο εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα δεν θα έπαιρνε τίποτα. Επειδή όμω είναι στη Γερμανία, ας πούμε στο εξωτερικό παίρνει τα 190 ευρώ και υπάρχουν χώρες που λένε ότι αν παίρνει επίδομα τέκνου σε άλλη χώρα σε εμάς δεν θα πάρει τίποτα. Η Γερμανία τα 190 ευρώ να τα δίνει σύνολο σε σένα και όχι 100 ε, εμείς και 90 Γερμανία. Και υπάρχει μια χώρα που από ό,τι ξέρω μάλιστα φορολογείται το επίδομα τέκνου. Αυτό είναι ε, κατά της ευρωπαϊκής Δημοτησίας, είναι λάθος, πρέπει να το ελέγξουμε. Σας λέω, το θέμα δεν είναι να ονοματίζουμε τις χώρες, ότι μία χώρα είναι καλή, άλλη είναι κακή. Εγώ απλά θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει πρόβλημα ο συνάδελφος, ο παρακαθήμενος, ε, είπε στοιχεία. Στην Γερμανία μιλάμε για 500 εκατομμύρια ε, το χρόνο ε, ή 1,5 δις νομίζω. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να αναπροσαρμόζουν τα επιδόματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι αναγκασμένα τα κράτη να παραμένουν στους κανόνες. Δεν υπάρχει αναπροσαρμογή, δυνατότητα αναπροσαρμογής. Αυτή είναι και η άποψη της ε, ε, ενεργεία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και το λέω αυτό και απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ευχαριστώ κυρία Σόιντροβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να ε, τραβήξω προς το τη συζήτηση, αλλά είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Μια έκθεση που μπορεί να φαίνεται κάπως τεχνική, μια παρατήρηση που να έχει τεχνικό χαρακτήρα αλλά τελικά μας οδηγεί στην εξέταση θεμελιωδών ζητημάτων. Το μπορεί να υπάρχει ζωή και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω καταλαβαίνω τα επιχειρήματα των συναδέλφων από τη Γερμανία και από την Αυστρία, γιατί αυτό έχει να κάνει και με εργαζομένου από την Τσεχία που εργάζονται είτε στην Αυστρία είτε στην ε, Γερμανία. Η πρόταση ξέρουμε, γιατί η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν ικανοποιητική, προέρχεται από τις ε, απαιτήσει του Ηνωμένου Βασιλείου ενώπιση του Brexit. Εν πάση περιπτώσει γίνεται λόγος για περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη που όμως μπορεί να μας οδηγήσει σε εντάσεις. Και θέλω τα πράγματα να τα κοιτάξουμε με ηρεμία και ψυχραιμία. Ο κύριος Γκέρικε μας είπε ότι 200.000 παιδιά εκτός Γερμανίας εισπράττουν κοινωνικά επιδόματα. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σούλτσε ότι στο πλαίσιο των φορολογικών σας υποχρεώσεων δεν θέλετε να επιδοτείτε τα επιδόματα άλλων. Αλλά εάν κάποιος πήγαινε να εργαστεί στην Τσεχία θα συνέβαλε με τις ε, φορολογικές υποχρεώσεις του, την εισφορά τη φορολογική σε όλα τα συστήματα, το εκπαιδευτικό, το φορολογικό, το ε, ασφαλιστικό και το καθεξής. Επομένως, το ότι ένα μέρος των ποσών που συλλέγονται με τους φόρους ωφελεί μια οικογένεια είναι πιστεύω σωστό. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξουμε την έννοια της ε, δικαιοσύνης και τις ισότιμης κατανομής. Και πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, άλλωστε έχω καταθέσει και τις σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή, ο κύριος Κορέλ, αν θέλει να σχολιάσει. Όχι. Και δίνω το λόγο στον κύριο Μπαλάς. Ο κύριος Κυρέλ φαίνεται προτιμά να με αφήσει εμένα να βγάλω, να διατυπώσω τα συμπεράσματα. Δεν θέλω λοιπόν να καθυστερήσω περισσότερο τις συζητήσεις γιατί είπα αρκετά στην αρχή. Θέλω να πω μόνο μια προκατακτική παρατήρηση εν παρόδο ότι βλέπουμε μια κάποια αντίφαση μεταξύ ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης, διακίνησης για τους εργαζομένους που ταυτόχρονα όμως δεν απάλλαξε ε, κανέναν από την ε, αντιπαράθεση για προς όφελος του συντονισμού μεταξύ των διαφορών κοινωνικών συστημάτων γιατί βλέπουμε τώρα σε αυτή τη φάση ότι ένας χώρος κινητικότητας σχεδόν απόλυτης κινητικότητας έρχεται σε σύγκρουση με το γεγονός ότι δεν έχουν αναρμονιστεί οι κανόνες. Εμάς δεν είναι δουλειά μας βέβαια αυτό. Εμείς πρέπει να δώσουμε απαντήσεις βέβαια. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο στο μέλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με περαιτέρω εναρμόνιση στους διαφόρους τομείς των κοινωνικών συστημάτων. Αυτό άλλωστε το καταδεικνύει και η σημερινή μας συζήτηση. Τώρα πάνω σε ποια αρχή θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Καταρχάς, η πιο σημαντική αρχή, και είμαστε Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, η πιο σημαντική λοιπόν αρχή είναι ότι η κινητικότητα την οποία επιθυμούμε των εργαζομένων θα πρέπει να βαδίζει παράλληλα με την προστασία αυτών των εργαζομένων. Λέει η κυρία Βέμπερ ότι έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Όντως, φυσιολογικό είναι άλλωστε. Αυτό σημαίνει και δημοκρατία. Ταυτόχρονα ωστόσο γνωρίζουμε ότι μεταξύ των αξιών του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ήταν και το ότι επιδιώκει ταυτόχρονα την κινητικότητα και τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας. Τι να κάνουμε. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορεί ο εργαζόμενος να ε, ωφελείται των δικαιωμάτων για τα οποία εργάζεται. Αυτονόητο μην έχει κανεί την εντύπωση, μην περιγράφει κανεί τα κοινωνικά συστήματα σαν να έρχονται να δίνονται οφειλήματα δωρεάν. Είναι ανταποδοτικά τα συστήματα. Έχουν διαφορετικούς ε, μισθούς, διαφοροποιημένε αμοιβέ και αντίστοιχα δικαιώματα, αλλά και με βάση την ε, ε, φορολογική εισφορά, δηλαδή την κάλυψη από τον εθνικό προπολογισμό, πάλι είναι διαφοροποιημένη η διάθεση των ωφελημάτων, δηλαδή δεν, δεν παίρνει κανεί ωφέλη, ευεργετήματα ή επιδόματα χωρί να τα δικαιούται. Αυτό πρέπει να μπορεί να ελέγχεται, ναι. Αλλά εάν κοιτάξουμε τώρα τις προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι τα κοινωνικά δικαιώματα που προσφέρει αυτή η πρόταση υπολείπονται πολύ των δικαιωμάτων που έχουμε εξασφαλίσει σε σχέση με το εργατικό δίκαιο. Ε, τρεις μήνες ε, ή έξι μήνες για το επίδομα ανεργίας μπορεί να φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες εξασφαλίζεται κάλυψη με επίδομα ανεργίας για τον άνεργο για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών. Μην τα λησμονούμε αυτά, πρέπει να τα κοιτάμε όλα. Επίσης, καταπολέμηση τη απάτη του εργοδότη, γιατί συνήθως περί αυτής πρόκειται, Πολύ συχνά είναι η απάτη προερχόμενη από τον εργοδότη, όχι από τον εργαζόμενο. Πρόσφατες άλλωστε μελέτες δείχνουν ότι είναι πολύ χαμηλότερα τα ποσοστά απατών από τους εργαζομένους. Και αυτό δείχνει τι, ότι ο εργαζόμενος Ευρωπαίος του Βορρά, του Νότου, της Ανατολής, της Δύσης, έχει τα ίδια δικαιώματα και ανάγκε. Το να λέει κανεί, κανεί δεν το πει βέβαια εδώ, αλλά περιπτώσει ότι ε, θα μπορούσαμε και να ανεχθούμε μια κοινωνική απάτη γιατί θα ήταν απλούστερο το σύστημα, λιγότερο γραφειοκρατικό, ουσιαστικά σημαίνει ότι εκθέτουμε τον εργαζόμενο σε παραβέστη δικαιωμάτων, σε ε, επισφαλείς θέσεις σε μη εξασφάλιση δικαιωμάτων που θα είχε στη χώρα προελεύσεως, στη χώρα καταγωγής και αυτό σας λέω είναι αντίθετο με τα δικαιώματα ουδήποτε εργαζομένου είτε είναι από τη Βόρεια ή την Νότια ή την Ανατολική ή τη Δυτική Ευρώπη ή και την Κεντρική. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε και ποια είναι τα οικονομικά ε, διακυβεύματα, τα πολύ σημαντικά. Βεβαίω δεν έχω καμιά αντίρρηση να τα συζητήσουμε. Θα σα πω λοιπόν το εξή. Κοινωνικά επιδόματα. Πέραν αυτών όμως, ιδιαίτερα προβλήματα και ανισορροπία για, για πολλές χώρες το ζήτημα της διασυνοριακής εργασίας. Όπως έχει τώρα το σύστημα της διασυνοριακής εργασίας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Ξέρετε ότι είναι ένα σύστημα με ανταπόδοση. Δισεκατομμύρια κοστίζει σε ορισμένα κοινωνικά συστήματα, ενώ κάποια άλλα εποφελούνται κάποια δισεκατομμύρια από τη δουλειά των υπερσυνοριακών εργαζομένων με το τωρινό σύστημα υπερσυνοριακής εργασίας ή διασυνοριακής εργασίας. Εδώ είναι τα προβλήματα που έχουμε. Εδώ είναι το οικονομικό διακύβευμα σε σχέση με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και βεβαίως άκουσα με μεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις και παρεμβάσεις που ζητούν περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων ε, για την διασυνοριακή απασχόληση. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλιστούν ουσιαστικά δικαιώματα για τον διασυνοριακό εργαζόμενο που έχει καταβάλει τις εισφορές του, που πρέπει να έχει δικαίωμα στην κατάρτιση, που πρέπει να έχει το δικαίωμα της νομικής αρρωγής χωρίς να βρίσκεται σε υποδέστερη ή πιο αδύναμη θέση. Και ναι, σήμερα μιλήσαμε πολύ για την δυνατότητα της προσαρμογής που δεν έχει γύρει η Επιτροπή γιατί δεν είναι στην πρότασή της των οικογενειακών επιδομάτων. Αλλά σε όρους οικονομικούς είναι πολύ πιο περιορισμένος ο αντίκτυπός τους από αυτό που εγείρω εγώ εδώ, δηλαδή επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη διανοσυνοριακή εργασία. Κύριε Σούλτσε αλλά και άλλοι συνάδελφοι που εγείρονται το θέμα αυτό, σας διαβεβαιώνω. Θα το συζητήσουμε, θα το ανοίξουμε το θέμα δεν πρόκειται να ε, σκουπίσω κάτω από το χαλί αυτά ή να ε, απορρίψω εκ προημίου ή οδήποτε ζήτημα ανησυχία. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι αυτό ο κίνδυνος για την ισορροπία των κοινωνικών μα συστημάτων. Πρώτον. Και επίσης θα πρέπει να πω κυρία Πρόεδρε, το είπε ο κύριος Σούλτσε πολύ σωστά, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και γιατί διότι χρειάζεται μια γενική συμφωνία. Εάν θέλουμε αυτή τη γενική συμφωνία θα πρέπει ο καθένας να δεχθεί είτε είναι από την Ανατολική, τη Δυτική, τη Βόρεια, τη Νότια Ευρώπη και την Κεντρική να μην κερδίζει πάντα ή να χάσει λίγο γιατί θα ξέρει ότι θα κερδίσει κάπου αλλού. Και ξέρουμε ότι είναι κακό να εμένουμε σε κάποιες θέσεις. Ο κύριος Κρίστενσεν, για τον οποίο τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση και ιδιαίτερα για τα λόγια που χρησιμοποίησε, γιατί ξέρω ότι ε, χρησιμοποίησε, ε, χρειάστηκε πολύ πολιτικό θάρρος για να μιλήσει όπως μίλησε. Αλλά είναι το παράδειγμα, πιστεύω. Το παράδειγμα που θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε και θα πρέπει να πούμε τι είναι το πιο σημαντικό για μας σήμερα. Και άρα να πούμε να εδώ μπορώ να περιορίσω τις απαιτήσει μου γιατί θα κερδίσω στο άλλο που είναι πιο σημαντικό. Στους σκιώδεις ηγητές λοιπόν θα παρακαλέ, τους ηγητές λοιπόν θα τους παρακαλέσω να κάνουν μια διαφοροποίηση μεταξύ της συλλογική θέση της ομάδας τους, την οποία εκφράζουμε στη συζήτηση αυτή, και την εθνική ή και προσωπική τους θέση που είναι κάτι διαφορετικό θεωρώ. Αυτά. Έτσι ξεκινάμε τη δουλειά. Είναι ικανοί όλοι οι συναδελφοί, πολύ ικανοί και με μεγάλη χαρά προσλέπω στη συνεργασία μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you for this. Σας ε, ευχαριστώ πολύ ε, και θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής στις 23 Μάλλον το είχα, είχαμε την παρουσίαση στις 23 Μαρτίου πέρυσι και τώρα ε, βαδίζουμε προς ε, έγκριση στις 19 Ιουνίου. Τουλάχιστον αυτό είναι το πρόγραμμα. Έχουν γίνει πάρα πολλές ε, συζητήσεις και πολύ σκληρή δουλειά κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση για το γεγονός ότι ήρθατε και θα επανέλθουμε ε, εν ευθέτω χρόνο. Η έγκριση στην Επιτροπή προβλέπεται για τις 19 ε, Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ και η επόμενη συνάντησή μας σε αυτή την Επιτροπή είναι ε, στις 21 και 22 Μαρτίου Άρα δηλαδή θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και που ε, λάβατε μέρος σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.